ελήψη αντιρρήσεων μπορώ να θεωρήσω ότι η μέρηση διάταξη γίνεται δεκτή. Σας πενθυμίζω τις αποφάσεις των συντονιστών στις 3 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Αποφασίστηκε καταρχήν να ζητήσουμε βάσει του άρθρου 54 η Επιτροπή μας θα συμμετάσχει στην εκπόνηση της έκθεσης του, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής δεν έχει ακόμα ε, προσδιοριστεί, αλλά θα προέρχεται από την ομάδα των σοσιαλιστών. Δεν ξέρετε ακόμα. Όχι, εντάξει. Επίσης, μία γνωμοδότηση στην έκθεση ΑΦΕΤ και ΕΦΚΟ για τις θεσμικές και πολιτικές ε, πτυχές μιας κοινή πολιτικής, ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας μετά την συνδίκη της αγοράς. Οι συντονιστές έχουν αποφασίσει να αποδώσουν αυτή την έκθεση στον Πρόεδρο, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφοι. Επίσης, έκθεση της Επιτρόπης αλληλεγγύη για τη διαχείριση των αλληλευτικών στόλων στις πιο απομεμακρυσμένες περιοχές ο εισηγητής θα πρόκειται από την ομάδα του ΕΛΚ. Ο κύριος Φερνάντε δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος από τις τάξεις του ΕΛΚ. Όχι ακόμα. Απόφαση για την ε, παροχή γνωμοδότησης στην Επιτροπή της ΑΦΚΟ για το θεσμικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής έρχεται από την ομάδα του ΕΛΚ γνωμοδότησε επίσης για την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών σε σχέση με την πολιτική και ασφάλειας και άμυνας, την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας και εδώ δεν υπήρχε κανένα <clears throat> υποψήφιος και οι συντονιστέ ε, έδωσαν αυτή την έκθεση στον πρόεδρο της Επιτροπής μα, επίση, προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλο της θητείας για το 2017 η έκθεση αυτή θα αποδοθεί στην ομάδα των Πρασίνων, για το 2018 στην ομάδα ECR, 2019 στο ΕΛΚ και 2020 για τους σοσιαλιστές. Και επίσης αποφασίστηκε ο κύριος Σίντζακ Ταραντ να είναι ο εισηγητής για, τις, για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού για, τα έτη, για το έτος 2017. Αποφασίστηκε επίσης η συμμετοχή στην ομάδα εργασία για την χρηματοδοτική αρρωγή θα πρέπει να αποφασιστεί από τι πολιτικέ ομάδε για να τηρηθούν οι απαραίτητε ισορροπίε και επίση αποφασίσαμε να μην εγείρουμε καμία αντίρρηση στην ε, συνέχιση του ειδικού εμπειρογνώμονο στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου στην Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτέ οι αποφασίε των συντονιστών 3 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο και απλώς τις έφερα και πάλι στη γνώση σας. Έρχομαι στα πρακτικά της ε, συνδιάσκεψης που έλαβε χώρα υπό Ολλανδική Προεδρία στο Άμστερνταμ στις 28 Ιανουαρίου με αντικείμενο τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Προεδρία των Κατοχωρών θεώρησε ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινή διαδικασία προβληματισμού για τις ε, συνθήκες κάτω από τις οποίες συζητούμε τα σχέδια προϋπολογισμών, για τις συνθήκες με τις οποίες διαμορφώνεται το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η ενδεχόμενη αναθεώρησή του. Η Προεδρία λοιπόν, η οποία μας υπέδεχτη στο Άμστερνταμ, τόνισε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όταν αναδύονται συνθήκες κρίσης, γιατί το πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο θέτει σε ένα πολύ στενό το δημοσιονομικό πλαίσιο και υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο ευκαμψίας. Το πρωί της ε, ημέρας εκείνης υπήρξε μια παρουσία προσωπικότητων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ίδιο ήμουν παρόν από την Επιτροπή Προπολογισμών και πολλοί από εμά με ύψιλον ήταν παρόντε. Η Αϊντα Κουάρντα Σαβάλ, ο Ζουαν Μανουέλ Φερνάντε, κ. Λεβαντόφσκι και κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Το πρωί χωριστήκαμε σε ομάδες εργαστηρίου το πρώτο εργαστήριο, το πρώτο ατέλειε προσπάθησε να καθορίσει τα χαρακτηριστικά αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ένα ιδεατό προϋπολογισμό. το δεύτερο ατελείο αφορούσε τα θέματα χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, παρουσία του Μάριο Μόντι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος τη ομάδα υψηλού επίπεδου. Ένα τρίτο ασχολήθηκε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων μας στον προϋπολογισμό και ιδίω κάτω από έκτακτες συνθήκες. Και το τέταρτο ατέλειο αφορούσε τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Τόσο για τον ενιάυσιο προϋπολογισμό, όσο και για τα πολιετή πλαίσια και για τις τροπολογίες που κατατίθενται στον ε, ετήσιο προϋπολογισμό. Μετά λοιπόν από αυτά τα τέσσερα πρωινά έλαβε χώρα η Σύνοδος Ολομέλειας της συνδιάσκεψης το απόγευμα. Με παρούσα την αντιπρόεδρο της Επιτροπής και αρμόδια του προϋπολογισμού την κυρία Κρυσταλίνα Τζόζεβα, η οποία με μεγάλη πεποίθηση και ενθουσιασμό αντιμετώπισε τα γενικά ζητήματα του προβληματισμού μας και προσπαθήσαμε να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα στην τελική συνεδρίαση το απόγευμα της ίδιας αυτής μέρας και τα συμπεράσματα αυτά συνοψίζονται σε δέκα σημεία. Πρώτον, θα πρέπει οι πολιτικές του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να διέπονται από την ανάγκη παροχής <clears throat> ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας. Είναι γεγονό ότι τα περισσότερα κονδύλια του ευρωπαϊκού προπολογισμού έρχονται από τα κράτη-μέλη, γιατί είναι κάτω από 10% τα ποσά που προέρχονται από τα τελωνιακού δασμούς και όσο προχωρούμε σε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών θα εκμηδενιστούν. Τα κράτη-μέλη φυσικά δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και 80% του προπολογισμού μα επανέρχεται στα κράτη-μέλη ως ε, κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, διαρθρωτικών ταμείων, κοινή αγροτική πολιτικής και εδώ υπάρχει η απέτηση να εξασφαλίσουμε ότι πρόρχεται από την διαδικασία αυτή και κάποια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. <clears throat> Δεύτερο πόρισμα θα πρέπει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να διαμορφώνεται με τρόπο δημοκρατικό και διάφανο. Με άλλα λόγια, να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναγνώσιμος από τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάθε εβδομάδα που γυρίζω στην εκλογική μου περιφέρεια έχω πολλές δυσκολίες να πράξω κάτι τέτοιο. <clears throat> Ιδίω σήμερα που έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, έχουμε καταστάσεις κρίσης, έχουμε ειδικά εργαλεία και διευκολύνσεις που πρέπει να επινοήσουμε και όλα αυτά η διευκολύνση του προπολογισμού, τα καταπιστεύματα, οι ειδικές, τα ειδικά κονδύλια για τη μετανάστευση και την Τουρκία. Πώς ακριβώς λοιπόν μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε πιο σαφή και πιο αναγνώσιμα από τους πολίτες μας. Τρίτο διδάγμα. Δεν θα πρέπει να σωρεύουμε πρόσθετους φόρους και επιβαρύνσεις για να έχουμε περισσότερους ίδιους πόρους. Με άλλα λόγια, αν <clears throat> δημιουργηθεί κάποιος νέος πόρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό δεν θα πρέπει να βαρύνει επιπλέον τους ε, φορολογούμενους και να προσθέσουμε ένα ευρωπαϊκό φόρο στους τοπικούς και εθνικούς φόρους. <clears throat> Αν λοιπόν αύριο θεσπιστούν ευρωπαϊκοί φόροι οι οποίοι θα ψηφιστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνεισφορές οι οποίες πληρώνονται από τους πολίτες στο εθνικό ή τοπικό επίπεδο να μειωθούν αντιστοίχω. Τέταρτο δίδαγμα. Χρειαζόμαστε να είναι επαρκής η προσθεμένη αξία όπως είπαμε προηγουμένως και η προσθέμενη αυτή αξία θα πρέπει να έχει ένα ευέλικτο χαρακτήρα. Όταν χρειαζόμαστε λοιπόν να ανταποκριθούμε άμεσα σε ε, αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν επιγόντως θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα ευελιξίας. Πέμπτον, χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση για οποιαδήποτε τροποποίηση στα έσοδα και τις δαπάνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνολική εικόνα και του τομέα δαπανών αλλά και του τομέα των εσόδων. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια άμεση σύνδεση μεταξύ του έργου μας για τις δαπάνες και του έργου μας για τα έσοδα. Έκτο δίδαγμα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία όταν ξεκινάμε τη συζήτηση και τον προβληματισμό για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, τα ανώτατα όρια των πόρων μας δεν θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται πλήρως στα διάφορα προγράμματα με προσδιορισμό ανακατηγορία θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο το οποίο θα είναι αρκετά ευρύ ώστε να μπορούμε να έχουμε πραγματική ευελιξία στη χρήση του προπολογισμού. Έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιον μας την κρίση του προσφυγικού και αυτό έκανε ανάγλυφο το πόσο δύσκολο είναι να έχουμε πόρους ελεύθερους όταν παρουσιαστούν τέτοιες κρίσεις. Έβδομο, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο συχνά και ευρύτερα τα εύκαμπτα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία βασίζονται σε μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Αυτό αφορά τη μόχλευση η οποία μπορεί να προκύψει, την χρήση του μέσου ευελιξίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων επίσης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. 8. <clears throat> Θα πρέπει η σωστή χρήση όλων αυτών των κονδυλίων να είναι κάτι το εφικτό, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι δαπάνες μας προσφέρουν την απαραίτητη προσθέμενη αξία και το πράττουν με τρόπο πιο είναι προς τους τεθειμένους στόχους. Ένα το στοιχείο, ένα το δίδαγμα και δεν έχει αυτό πολύ εύκολο. Έχουμε τονίσει πάρα πολύ την έννοια της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να καθορίσουμε με σαφήνεια τι ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή υποστημένη αξία. Και δέκατον και τελευταίο δίδαγμα, μέσα στα πλαίσια των ε, επερχομένων <clears throat> πολιετών δημοσιονομικών πλαίσιων θα πρέπει να διαπραγματευτούμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους και να προσδιορίσουμε την υποστημένη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει να κάνει με τους στόχους αυτούς και να κινητοποιήσουμε τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Συνοπτικά λοιπόν, αυτά είναι τα, αν θέλετε, τα συνοπτικά πρακτικά αυτής της συνδιάσκεψης του Άμστερνταμ. Αλλά φυσικά θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σας σχόλια, ιδίως από αυτούς οι οποίοι ήταν παρόντες στην συνδιάσκεψη αυτή. Κυρία Γουαρδιά Ζεράλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συνοψίσατε τέλεια νομίζω τα θέματα που εξετάστηκαν σε αυτή τη διάσκεψη. Αλλά σύνοψη είναι. Και όσοι συμμετείχαμε στις ομάδες εργασίας παρακολουθήσαμε συζητήσεις ενδιαφέρουσες όπου σε κάποιες είδαμε προς τα που κάποιοι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προσανατολίζονταν. Κάτι που με παραξένεψε στη διάσκεψη στο γενικό θέμα είναι ότι κανείς δεν μίλησε για την ανθεώρηση του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου. Δηλαδή είχε επικεντρωθεί η συζήτηση σε μια απλή και χαλαρή συζήτηση για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί φάνηκε ότι η πλειοψηφία το θεωρούσε δεδομένο αυτό το πλαίσιο, εγκεκριμένο μέχρι το 2020 και ότι η συζήτηση αφορούσε το μέλλον. Αυτό με ανησυχεί όμως, επειδή το τωρινό πλαίσιο χρειάζεται ακόμα πολλή συζήτηση. Εγώ ήμουνα στην ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με τις νέες προτεραιότητες και τη χρηματοδότησή τους. Κυρίως επικεντρωθήκαμε στην ευελιξία στα πλαίσια του πλαισίου. Κανείς ας πούμε δεν είπε αν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα λιγότερα χρήματα, αν το τωρινό πλαίσιο επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, τις κρίσεις και τα καταπηγόντα που έχουμε μπροστά μας, απλά και μόνο χαλαρά μιλήσαμε για την ευελιξία. Και να λέγει ότι όσοι πήραμε μέρος, συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Δεν φτάσαμε όμως στο ψητό τι είδος ευελιξίας χρειαζόμαστε, δηλαδή να αφαιρέσουμε από κάποια προγράμματα και να τα βάλουμε σε άλλα πιο επίγοντα. Ή τέλο πάντων, αν περισσότερη ευελιξία σημαίνει ότι θα έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για 7 χρόνια και μετά προσαρμοζόμαστε σε ό,τι προκύψει. Χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να αφαιρέσουμε κονδύλια από υπάρχοντα προγράμματα. Προκατακτική λοιπόν συζήτηση, δεν είχαμε χρόνο να ψηφίσουμε σε λεπτομέρειες και βέβαια δεν κάναμε διαπραγματεύσεις για το μέλλον του νομισονομικού πλαισίου. Κάτι άλλο που με ανησύχησε, τουλάχιστον στη δικιά μου ομάδα εργασία, ήταν η επιμονή για τα εργαλεία, το οικονομικά στον προπολογισμό. Ανέκυψε επανειλημμένο το μεγαλείο του σχεδίου επενδύσεων Juncker ως φάρμακο ευρωπαϊκή. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος αποτελεσματικός για να δαπανηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, οπότε η λύση για το μέλλον ήταν το να μετατρέψουμε ας πούμε τους προπολογισμούς μας και το δημοσιονομικό πλαίσιο σε κάτι το οποίο θα είναι γραμμές για την δημιουργία υποδομών και εργαλείων σύμφωνα με το σχέδιο Juncker. Αλλά με ανησυχεί μεταξύ άλλων και για το γεγονό ότι μόλι ξεκίνησε αυτό το σχέδιο Juncker και δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι καλό για τι επενδύσει ή όχι ανεξάρτητα από το αν θα είναι αποτελεσματικό ή όχι το σχέδιο του Γιούνκερ. το θέμα είναι ότι ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από εργαλεία χρηματοοικονομικά. Επανειλημμένω, τα συζητήσαμε σε αυτά εδώ στην Επιτροπή μα και πάντοτε καταστήσαμε σαφέ και το πάμε και στη συζήτηση για το σχέδιο Γιούνκερ ότι αυτά τα εργαλεία ισχύουν και αξίζουν για κάποιε πολιτικέ για κάποιε περιπτώσει και για κάποιου τομεί. Η αγορά δηλαδή μόνη τη δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει, αλλά δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι εδώ χρηματοδοτούμε αποκλειστικά μέσω επιδοτήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε τα επόμενα χρόνια λοιπόν και νομίζω ότι είναι αρκετά επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή είναι η θέση που έχουμε εμείς στην σοσιαλιστική ομάδα. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε ένα προπολογισμό αποκλειστικά στην ουσία προπολογισμό χρηματοοικονομικών εργαλείων. Κάθε πρόγραμμα, κάθε κατάσταση στην αγορά, κάθε περίπτωση χρειάζεται διαφορετικά εργαλεία. Άλλα θα στρέφονται προ την αγορά, άλλα θα αποτελούνται από επιδοτήσεις, ας πούμε στη Γεωργία. Δεν ξέρω πώ μπορούμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία. Έχουμε την ΚΑΠ και βεβαίω υπάρχουν και τομεί και προγράμματα που θα μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα εργαλεία. Μιλάω για αυτά επειδή στην ομάδα εργασίας που συμμετείχα το συζητήσαμε ευρέως και επαγγελμένα ακουγόταν ως παράδειγμα το σχέδιο επενδύσεων του Juncker και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελήσει πανάκια για όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Πάντως, νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η διάσκεψη για την αλήθεια ότι είχαμε ένα διαφορετικό περιβάλλον συζητήσεων από αυτό που έχουμε Συνήθω. Είχαμε εκπροσώπου κυβερνήσεων, κοινοβουλίων, υπουργείων, γεωργία, ελεκτικών συνεδρίων. Είχαμε έτσι μια χαλαρή και ήρεμη συζήτηση για να αναζητούσουμε έτσι καινοτόμους τρόπους εξέτασης του μέλλοντος. Υπάρχουν βέβαια πολλοί αποκλίνουσες απόψεις για το επόμενο δούπου και στην αναθεώρηση υπάρχουν ακόμα πολλά που θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω κάποια πράγματα στην εισαγωγή. Πιστεύω και εγώ ότι η διάσκεψη που είχε οργανωθεί πολύ καλά και που είχε και πολλούς ε, παρόντες ε, ασχολιόταν κυρίως με το μέλλον, ενώ νομίζω ότι αυτό μας πιέζει περισσότερο είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα συναντήσουμε κάποια προβλήματα στον προϋπολογισμό πριν το 2018 ή το 2019 και θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά την ουσία, το μάντρα, το σύνθημα μας σήμερα, είναι να έχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αλλά νομίζω ότι για πολλούς ε, από τους ε, συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτό ισοδυναμεί με ε, κεντρική διαχείριση αλλά αυτό είναι μια χοντροειδής απλοποίηση. διότι όλα έχουν να κάνουν με την ε, στάση μας απέναντι στην Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά το λεξιλόγιο της ε, διάσκεψης ε, ήταν φορτωμένο με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. αναφέρθηκε η διαφάνεια, ο καλύτερος έλεγχος ε, του προϋπολογισμού, η ε, ευελιξία και η τάση να ε, προχωράμε από στην μόχλευση. Εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο Juncker θα είναι λειτουργικό και θα ωφελήσει το, τη Βόρεια Ευρώπη και όχι απαραίτητα τις χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση ε, στην ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αποκλειστικά με τη φιλοσοφία αντικατάσταση ε, των χορηγιών ε, από επενδύσει μόχλευσης. Ε, Πάντω και εγώ την ίδια εντύπωση έχω για τη διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Οντή, ήσασταν παρούσα και εσείς, έτσι δεν είναι. Δυστυχώς όχι. Αλλά να συνεχίσω κι εγώ και ενδεχομένως να επιβεβαιώσω τι παρατηρήσει αυτών που ήταν παρόντε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις ε, που έγιναν. Αναφερθήκατε στην ε, ανάγκη ορισμού της προστιθέμενης αξίας ε, και αυτό ισχύει για το σχέδιο επενδύσεων. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή αν πληρούνται τα κριτήρια. Και δεν ε, έχει αποδειχθεί ακόμα ότι η μόχλευση είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να εξετάσουμε τον προϋπολογισμό και να δούμε πού ε, θα χρειαστούν χορηγίες και πού θα χρειαστεί η μόχλευση. Θα πρέπει να ε, μην ξεχάσουμε το θέμα ε, των επιδοτήσεων. Πέρα από αυτό όμως όσον αφορά την έννοια της προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει να εξετάσουμε τον προϋπολογισμό και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και είναι ενδιαφέρον το ότι αναφέρθηκε τόσο συχνά. Και η τελευταία μου παρατήρηση όσον αφορά τα δέκα συμπεράσματα και τη διάγνωση των προβλημάτων. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς τη διάγνωση. το, η λύση είναι το πρόβλημα. Όταν λοιπόν μιλάμε για ευελιξία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της, ε, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σταθερότητα και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή τη σταθερότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμακετ που είναι παρούσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν άκουσα όλα αυτά που είπαν ε, οι προαλαλήσαντες γιατί ήθελα λίγο καθυστερημένη. Προσπαθώ να είμαι σύντομη γιατί τα περισσότερα έχουν ελεγχθεί ήδη. Αυτό το οποίο εγώ βρίσκω πολύ εκπληκτικό είναι ότι όλοι μιλάνε για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κανείς δεν μιλάει για την αναθεώρηση στη μέση του δρόμου του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Σαν να είμαστε σε άλλο πλανήτη. Δεύτερον, όπως είπε ο κύριος Λεβαντόφσκι και άλλοι, μιλάμε σαν να έχουμε το μαγικό ραβδάκι της προσθεμένης αξίας. Αλλά φοβάμαι ότι όπως είπε και η κυρία Οντή, δεν συμφωνούμε καν για το τι ακριβώς αποτελεί αυτή την προσθέμενη αξία. Γι' αυτό βρισκόμαστε μέσα σε μια ασάφεια και περισσότερο σε μαγικό ρεαλισμό παρά σε πραγματικότητα. Σαν παράδειγμα, ο κύριος Φερναντές στην επιτροπή που ήμασταν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αρχές του προϋπολογισμού οι οποίες να είναι οι αρχές της προτεραιότητας και μίλησε για αλληλεγγύη ο μόνος ο οποίος μίλησε για αλληλεγγύη βέβαια από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν. Θεώρησε ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι ένα κομμάτι του, των αρχών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν το λέγανε, δεν το είπαν και πολλοί άλλοι. Και κάποιο άλλο μαγικό ραβδάκι το οποίο αναφέρθηκε ήταν αυτό της ε, ευελιξίας. Μα και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι η ευελιξία είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να βρούμε πρόσθετα κονδύλια με τις ε, ευελιξίες, <clears throat> να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας, αλλά αυτό σημαίνει, όπως είπε και η κυρία Γουάδια Σαμπάλ, ότι θα είμαστε στην ανάγκη να έχουμε παγκόσμια κάποια προγράμματα τα οποία είναι λιγότερο προτεραιότητα στον ορίζοντα 2020 για να γεμίσουμε τρύπες αλλού. Υπενθυμίζω αυτά που είπε ο κύριος Μόντι. Είπε ότι η έννοια της ευελιξίας ήταν κάτι που ομόφωνα το αποδεχόντουσαν οι παρόντες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, στον εθνικό προϋπολογισμό, δεν αντιμετωπιζόταν το θέμα της ευελιξίας με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν ο ίδιος ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός μπορεί μερικές φορές να έχει ελλείμματα. Ίσως χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και λιγότερη ευελιξία στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό θέλω να πούν ίσως. Κόλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στις ε, συζητήσεις. Ωστόσο, μου άρεσαν κάποιες ε, παρεμβάσεις και της κυρίας Καβασβάλ και του κυρίου Λεβαντόφσκη εάν σωστά ερμηνεύω αυτό που άκουσα, Φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν είναι αυτό το θαυματουργό όπλο με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια συζητήσεων για το ΕΦΣΥ Είχαμε έναν ομιλητή που είδε επικριτικά το Ταμείο αυτό, ενώ όλοι οι άλλοι θεώρησαν ότι αποτελεί ε, θαυματουργό μέσο. Ίσως ε, στις επόμενες ε, συζητήσεις θα πρέπει να δούμε από πιο νωρίς επικριτικά το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς το αναφέρατε. Σημαντική είναι η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες μας ε, και δεν μπορώ να φανταστώ να αυξάνεται η διαφάνεια εάν ε, βάλουμε ένα σωρό χρήματα σε ταμεία και κάποιοι φορείς αποφασίζουν για την ε, κατανομή τους. Η διαφάνεια σημαίνει και έλεγχος των δαπανών. Και βέβαια τίθεται το θέμα πόσο ευέλικτος μπορεί να είναι ένας προϋπολογισμός. Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, ωστόσο να ρωτιέμαι πώς μπορούμε με άλλο τρόπο να έχουμε έναν κάποιο έλεγχο από πλευράς του Κοινοβουλίου. Στο μέλλον λοιπόν όταν θα μιλάμε για τέτοια προγράμματα σας παρακαλώ ας έχουμε επικοδομητική αλλά και επικριτική στάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να κάνω μερικά σύντομα σχόλια λέει κύριο Μπέργκερ. Δεν ισχύει ίσως το ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν συνεπαρμένη. Όχι αγωνιστήκαμε και διαπραγματευτήκαμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε ένα εξισορροπημένο πακέτο και αυτό είναι για μένα ένα είδος, είχαμε ένα μεγάλο πιλωτικό πρόγραμμα, το Ταμείο Επενδύσεων και κατά τα άλλα πήραμε κάποια κονδύλια από την, Επίτρο, από την πολιτική έρευνα και μεταφορών. Δεν ήταν καθόλου εύκολο και σας μίλησα για ένα πιλωτικό πρόγραμμα γιατί το ερώτημα αυτό είναι πραγματικά δικαιολογημένο. Αν λόγω της ιστορικής οικονομικής κατάστασης και της πολιτικής επιτοκίων είναι πράγματι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο ταμείο, επενδυτικό ταμείο. Στη δική μου εκλογική περιοχή, στα βόρεια του Αμβούργου, υπάρχει το σχέδιο για ένα αυτοκινητόδρομο με τέσσερις ε, λωρίδες που θα γίνει έξι και που είναι ένας δρόμος ο οποίος συνδέει το Αμβουργό με την ε, Σκανδιναβία. Αλλά οι εξαγωγές οι οποίες θα εξυπηρετήσει δεν έχουν πια τόσο μεγάλο νόημα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε ήδη εξεταστεί στο χρονικό διάστημα 2006-2013. Δεν έγινε από το μηδέν λοιπόν αυτό. Είχαμε ήδη ξεκινήσει με μια συμφωνία για ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την Κομισιόν για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Μάλλον τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συγγνώμη. Και αυτό ήταν ένα σχέδιο σύμπραξη ιδιωτικού και <clears throat> δημοσίου τομέα. Μισό ε, δημόσιο χρήμα, μισό ε, ιδιωτικά κονδύλια, τα οποία όμως ε, θα καλυπτόντουσαν με εγγύησει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα χρηματοδοτούνται με τα διόδια των φορτηγών. Αυτό, μπορούσε Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει λοιπόν πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα σχέδιο το οποίο είναι καθαρά δημόσιο. Βλέπουμε λοιπόν ποιε είναι οι δυνατότητες που μπορούν να δημιουργηθούν. Πρέπει να εξετάσουμε τέτοια παραδείγματα, αλλά έχει σημασία και το πώς θα λειτουργήσει ο προϋπολογισμός. Δεν μπορεί ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωση να λειτουργεί μόνο μέσα από χρηματο ε, χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης. Τίθεται και το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου. Και αυτό ισχύει <clears throat> και για όλα τα ταμεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί, παραδοσιακά το Ταμείο για την Αφρική και όλα αυτά τα έχουμε δεχτεί, αλλά τα έχουμε δεχτεί με μεγάλη δυσκολία γιατί με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά διαβρώνονται οι δυνατότητες ελέγχου και απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλα αυτά τα εξωτερικά ταμεία Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με θετικό τρόπο ώστε να δώσουν και πρόσθετα κονδύλια εκεί που χρειάζεται, αλλά εμείς έχουμε πολλά ερωτηματικά αυτή τη στιγμή. Και <clears throat> τίθεται και το θέμα του αν με τον τρόπο αυτό κατακαιρματίζουμε τον δημοσιονομικό χώρο Αν λοιπόν όταν χρησιμοποιούμε την ευελιξία με όλα τα κονδύλια ήδη στο μισό το πρώτο του χρόνου και μετά στο τελευταίο μισό δεν έχουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Και για να αντιμετωπίσουμε ανάγκες πρέπει να κάνουμε μεγάλες αναδιατάξεις στις κατηγορίες του προϋπολογισμού όπως είναι στην κατηγορία 4 όπου χρησιμοποιήθηκε μια διαδικασία ταχείας απόφασης για μια μεταφορά 9 ε, δισεκατομμυρίων. Και έχουμε επίσης και προγράμματα τα οποία έχουν ε, να κάνουν με την προενταξιακή βοήθεια και με την ε, πολιτική γειτονία, στα οποία έχουν αφαιρεθεί από τον προπολογισμό. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό έχουν ανατραπεί τελείως οι προτεραιότητες. Ίσως όμως θα πρέπει να έχουμε και μια πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε τον περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει πρέπει να θέσουμε το ερώτημα <clears throat> γιατί τα προγράμματα τα οποία έχουμε θεσπίσει για τη γειτονιά μας γιατί δεν έχουν λειτουργήσει ή τουλάχιστον τα αποτελέσματά τους δεν ήταν αυτά τα φιλόδοξα τα οποία θέλαμε και αν δει κανείς τώρα την κρίση με την ε, όξυνσή της, με τη μαζική μετανάστευση, τι μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν μετά από όλα αυτά. Και τι μπορούμε να συμπεράσουμε, να συμπεράνουμε. <clears throat> ότι αν δεν μπορέσουμε να υπάρξει μια πραγματικά ε, αναθεώρηση των ε, κονδυλίων στην κατηγορία 3 και 4, σκεφτείτε την Frontex, σκεφτείτε την ανάγκη προάσπισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας σκεφτούμε το τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να υπάρξει μια σταθεροποίηση των οικονομικών συνθήκων στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Όλα αυτά μας φέρνουν σε μια νέα κατάσταση που θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα εξασφαλίσουμε την σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν για μένα πολύ περισσότερες κοινέ ενέργειες, αλλιώς δεν χρειάζεται καν να συζητάμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενότητα. Και το Συμβούλιο πρέπει να ε, καταλάβει ορισμένα πράγματα. Ποτέ δεν είχαμε τόσες πολλές σωρευμένες κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε από τη μια μεριά τον Πούτιν, από την άλλη μεριά τον Τραμπ και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα τα οικονομικά του προπολογισμού μας. Χωρίς λοιπόν να υπάρξει μια δραστήρια αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα του θέματος της σταθεροποίησης του ευρώ. Άμα δεν κάνουμε τίποτα λοιπόν γιατί όλα είναι παρά υπερβολικά πολύπλοκα, δεν είναι θετικά τα πράγματα για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια επαναφορά στα εθνικά κράτη, στην κυριαρχία των εθνικών κρατών, όταν η πραγματικότητα μας δείχνει ότι αυτά τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση από μόνα τους να λύσουν κανένα πρόβλημα πια σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αλλιώς αυτά τα θέματα. Έχουμε την εξή λοιπόν το εξή δίλημα. Είτε θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αίτηση αναδιάταξη όλων αυτών, αν το Συμβούλιο λοιπόν τώρα δεν το δεχτεί αυτό το πράγμα, τότε θα πρέπει να γίνει σαφές και στα δύο αυτά τα θεσμικά όργανα ότι έχουν άλλα τρία έτη προϋπολογισμού μπροστά τους στο πολιετές πλαίσιο. Είτε θα κάνουμε μια πραγματική πρόοδο και θα ελέγξουμε πού υπάρχουν οι δυνατότητες εξοικονόμησης ή καλύτερης χρησιμοποίησης κονδυλίων. Αν μπορούμε λοιπόν να βρούμε αν οι προτεραιότητές μας είναι έγκυρες στο μέλλον, για το μέλλον ή όχι, ή όχι, και όποιος δεν δεχτεί να κάνει αυτή την άσκηση, αυτός αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Μόνο λοιπόν με το να έχουμε μια νέα δομή για ορισμένα θέματα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και εκεί είναι φανερό ότι στις κατηγορίες 3 και 4 είναι απαράγραπτη η, η αναδιάταξη του προϋπολογισμού, αλλιώς σε δύο χρόνια έτσι και αλλιώς θα έχουν τελειώσει όλα. Ευχαριστώ, κύριε Σταράν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Ήταν εφορίες που μας κάνουν να σκεφτούμε κάπως και λυπάμαι που δεν πήρα μέρος σε αυτές τις συναντήσεις. Δεν ξέρω πάντως αν αυτά που θα πω θα είναι είδος προειδοποίησης ή αν ακούγονται ως άποψη μάρτυρα. Κάθε φορά που μιλάμε για προστέμενη αξία θυμάμαι τον Μάρξ και την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό ακριβώς ως ορισμό της προσθεμένη αξίας. Euh, ναι, ευχαριστώ. Και τώρα νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξαναγίνει. Και... Ναι, ευχαριστώ. Ούτε και εγώ μπορούσα να πάω, αλλά άκουσα τι υπόθηκε ιδιαίτερα για το πλαίσιο. Να δούμε κατά πόσο ότι προβλήματα υπάρχουν, να δούμε μια έκθεση με στατιστικές και δεδομένα και μετά να υπολογίσουμε κατά πόσο αποδίδει ή όχι. Ποτέ δεν είπαμε ότι αυτό θα ήταν πανάκια. Ένα αυτό. Μετά. Αυτά που είπαμε στην διάσκεψη για το επόμενο πουδουπού. Νομίζω ότι εδώ σιγά σιγά βαδίζουμε από κρίση σε κρίση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια. Έχουμε προγράμματα με το Λίντερ για τη χώρα μου, ίσως και αλλού, που δεν έχουν δοθεί χρήματα ακόμα. Από ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι γίνεται με το τερνό δουπού και να μην συνεχίζουμε να πράττουμε σαν να συμβαίνει τίποτα, γιατί υπάρχει θέμα εδώ σταθερότητας και ελαστικότητας. Να το αντιμετωπίσουμε τώρα λοιπόν, διαφορετικά τα πράγματα δεν φαίνονται να, να είναι καλά τα επόμενα χρόνια. Προσβλέπω λοιπόν με χαρά στις αυρινές συζητήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρος. Ο κύριος Μακά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Και εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω τις δικές μου απόψεις σε σχέση με αυτό το γεγονός, αυτή την εκδήλωση, στην οποία εγώ δεν μπόρεσα δυστυχώς να είμαι παρόν. Και να σταθώ στο θέμα του Ταμείου Επενδύσεων Γιούνκερ. Όταν παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο από την Κομισιόν, ξέρουμε ότι ο, σχόλιο, ότι ο στόχος της ήταν να ξαναξεκινήσει η ευρωπαϊκή ατομηχανή, να υπάρξουν επενδύσεις σε τομείς όπου υπήρχε μεγάλη προσθέμενη αξία και μεγάλες αποδόσεις. Ο στόχος μας ήταν να υπάρξουν επενδύσεις σε τομείς όπου θα μπορούσε να ανακτήσει ο επενδυτής τα χρήματά του, αλλά συγχρόνως και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Δεν είχε νόημα να εφαρμοστεί σε τομείς όπου αυτό δεν θα γινόταν. Είναι απαραίτητο να έχουμε και μια αντιστάθμιση κινδύνων <clears throat> σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ αναρωτιόμουν πραγματικά τι είδου σχέδια θα μπορούσαν να παρουσιαστούν τα οποία δεν θα μπορούσαν να, να υλοποιηθούν αλλιώς. Και μόνο με το ΕΦΣΥ θα μπορούσε να γίνει. Αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν, εγώ είδα ότι ήταν παρόμοια με αυτά τα οποία χρειάστηκε εγώ να αντιμετωπίσω ως επικεφαλής μιας περιφερειακής αρχής. Γιατί λοιπόν να υπάρξει αυτή η απόσυρση κονδυλίων από το ορίζον 2020 και από άλλους τομείς και να τα επενδύσουμε σε άλλους τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς το FC έτσι κι αλλιώς. Επομένως τα σχέδια αυτά που παρουσιάστηκαν δεν ήταν τα κατάλληλα. <clears throat> θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το EFSI σε σχέση με την αρχική του σύλληψη. Δηλαδή να επενδυθούν χρήματα εκεί όπου κανένας άλλος επενδυτής δεν θέλει να μπει και να εξασφαλίσουμε τους κινδύνους αυτών των επενδύσεων. Ευχαριστώ, Λεωπρόεδρος θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα της, ε, του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Επενδύσεων Γιούγκερ. Αύριο ή μεθαύριο θα είμαι σε μια συνεδρίαση όπου θα προσπαθήσουμε να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα είδος απολογισμού για να δούμε αν η δέσμευση κονδυλίων και οι δανειοδοτήσεις και όλα αυτά συνάδει με τις ε, προϋποθέσεις που είχαμε θέσει για το ΕΦΣΙ. Ο κ. Κολμέλη, ένα τελευταίο σχόλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Γιατί μου πήρε το ψωμί από το στόμα ο κύριος ε, Μάνκα, κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στην απόκτηση συγκεκριμένων στοιχείων και λεπτομεριών για το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής το ΕΦΣΥ. Νομίζω ότι όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο όγκο χρηματοδότησης δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλο του προγράμματος για να δούμε ότι ενδεχομένω μπορεί να μην λειτουργήσει αυτό. Αυτά που είπε ο κύριο Μπέγκε με τον αυτοκινητόδρομο του Αμβούργου. Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν πράγματι ένα πρόσθετο σχέδιο ή αν ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να είχε γίνει και χωρίς τέτοια χρηματοδότηση. Μα τέτοια ερωτήματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι θα πρέπει να κατατήσουμε ένα ερωτηματολόγιο ώστε χωρίς τώρα να υπερφορτώσουμε την Κομισιόν να μας πούν πόσες αιτήσει έχουν υποβληθεί για το ΕΦΣΥ, πόσες εγκρίθηκαν, πόσες απορρίφθηκαν, με ποια κριτήρια, σε ποιο χρονικό ορίζοντα όλα αυτά, ώστε να έχουμε τουλάχιστον μια ιδέα για το τι γίνεται και κάποια συγκεκριμένα τα παραδείγματα. Θα γίνει αυτό, λέει ο πρόεδρος. Ωραία, προστεθεμένη αξία για ένα αυτοκινητόδρομο, στη Γερμανία αν καταβάλει τέλο πάντων την συμβολή της η Γερμανία στον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό και μετά αυτά τα χρήματα πάνε τέλο πάντων στον γερμανικό αυτοκινητόρμο, τότε αυτό είναι προς τα εξία. Θα δούμε πάντως πώς θα το προσεγγίσουμε όπως το παρουσίασε το θέμα κ. Σταράν και πολιτικά και ιστορικά. Ήταν πάντως ενδιαφέρουσα αυτή η διάσκεψη αναφυσβήτητα. Τώρα το θέμα είναι να δούμε τι συνέχεια θα της δοθεί. Πάντως έχω την εντύπωση εγώ ότι έχουμε ένα προπολογισμό που είναι κάπως αναχρονιστικός. Δηλαδή σχεδιάστηκε σε σχέση με τις τότε προσδοκίες όταν όμως έχουμε μια συγκεκριμένη, να κάνουμε μια συγκεκριμένη κρίση και οτιούνται οι πολίτες τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη τότε δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Και τώρα θα κάνω μια σύντομη σύνοψη αυτών που διαμήφθηκαν στην αποστολή που είχαμε 11 μέλη της ε, Επιτροπής μας 8 με 11 Φλεβάρι. Φρέσκα νέα λοιπόν, να δούμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Θα κλείσω εδώ το σημείο που αφορά την σύνοψη της διάσκεψης στο Άστερνταμ που διοργανώθηκε από την Ολλανδική Προεδρία 28 Γενάρη και να πέρασουμε σε ένα θέμα το οποίο αναφέραμε στο σεμινάριό μας πριν από ένα χρόνο πάντοτε επί της ίδιας προβληματικής για την Τουρκία η αποστολή αυτή της Επιτροπής μας πήγε η ομάδα μας εκεί, η Επιτροπή μας 8 με 10 και στις 11 Φλεβάρι είδαμε, εξετάσαμε μάλλον το πώς ακριβώς εφαρμόζονται και δαπανώνται αυτά τα κονδύλια σε αυτή τη φάση της προπροσχώρησης. Έχουμε αυτή τη δική φάση πριν από την προσχώρηση που αφορά τα έτη 2007 με 2013 για περίπου 5 δις ευρώ και μετά έχουμε ένα δεύτερο ειδικό εργαλείο προ-προσχώρησης, 14-20, γύρω στα 4,8 δις. Σημαντικά ποσά δηλαδή, τα οποία διατίθενται στην Τουρκία. Θα πρέπει να δούμε επίσης το πώς ακριβώς θα διοργανωθεί και η οικονομική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση των προσφύγων στην Τουρκία. Η αποστολή μας λοιπόν δούλεψε σκληρά, συμμετείχε σε συναντήσει, συνεδριάσει, στρογγυλέ τράπεζες, γεμάτα εργασία. Συναντήθηκε με γύρω στου 40 επισήμω συνομιλητέ, χωρί να απολογίσουμε τους άτυπα συνομιλούντε. Είχαμε εκπροσώπους από την Συρία, από τα κοινοβούλια τα γειτονικά, οργανώσεις, μη κυβερνητικέ, που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα συνομιλητέ με τις, με τους των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωτερικής δράσης, της Ευρωπαϊκή Τραπέζας Επενδύσεων και εκπροσώπων των χωρών μελών και επίσης υπηρεσιών που εκπροσωπούν πολλά κράτη-μέλη. Πήγαμε στην για την Δετάρτη για δύο επισκέψεις σε στρατόπεδα προσφύγων καταρχάς και μετά κάναμε μια επίσκεψη σε ένα σχολείο στον Γκάζι σχολείο της UNICEF που το έχτισε και το διαχείρισε η ίδια επειδή 9 στους 10 πρόσφυγες ε, έχουν ε, μοιραστεί σε διάφορες ε, κοινότητες μία εκ των οποίων είναι το Γκαζιαντέπ και πολύ συχνά ζουν έτσι σε πολύ αδίξω συνθήκες αυτή, η πρόσφυγες και προφανώ τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Είχαμε λοιπόν την επίσκεψη αυτή, έχουμε την πλήρη αναφορά της επίσκεψης, αλλά ήδη από τώρα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και να προκαταβάλουμε κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις και κάποια συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί οικονομικά για την προσχώρηση της ε, Τουρκία. 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Η Ευρωπαϊκή όμως Τράπεζα Επενδύσεων και αυτή θα παρενέβει στην ε, Τουρκία για περίπου 2 δι ετησίως. Η Ευρώπη παραμένει δεσμευμένη, δηλαδή θα παράσχει εργαλεία και κονδύλια και εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και εργαλεία επίσης ε, στήριξης της κοινωνίας των πολιτών τη Τουρκία, Η κατάσταση όμω όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων και οι κίνδυνοι που διατρέχει η Ευρώπη κάνουν την Ευρώπη να είναι κάπως διστακτική να ασκήσει δηλαδή κριτική προς την Τουρκία ιδιαίτερα για τα θέματα των ανθρωπινών ε, δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκρασης, της ελευθερίας του τύπου. Η Ευρώπη είναι παρούσα με γύρω 550 υπαλλήλου και εκπροσώπου κυρίως μέσω της ε, αντιπροσωπείας μας στην Άγκυρα. Έχουμε επίσης και διάφορες ΜΚΟ που λαμβάνουν τμήμα αυτών των κονδυλίων με άμεση διαχείριση. Έχουμε επίσης και κάποια εργαλεία όπως το Ταμείο ΕΚΟ και το Εργαλείο για τη Δημοκρατία και την Ειρήνη. Είναι σημαντική πρόκληση η υποδοχή των Σύριων προσφύγων. 2,5 εκατομμύρια περίπου είναι αυτοί που ζουν στην Τουρκία δηλαδή, αν προσθέσουμε και αυτούς που έρχονται από το Ιράκ ή το Αφγανιστάν και από το Ιράν, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι προσπάθειες που καταβάλουν οι τουρκικές αρχές για την υποδοχή αυτών των πληθυσμών. Και βλέπουμε ότι κάνουν ό,τι μπορούν οι οικογένειες που φιλοξενούνται εκεί φαίνεται να ζουν σε ικανοποιητικέ συνθήκες. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν βιβλιοθήκες για τα παιδιά, σχολικές υποδομές, ε, παντοπολία, σούπερ μάρκετ. Έχουμε μια υπηρεσία τουρκική που ασχολείται με την ε, διατροφή με την πιστική βοήθεια παγκοσμία. Έχουμε μια κάρτα η οποία τους παρέχεται για την διατροφή τους με 50 λίρες συν 35, 85 λίρες δηλαδή Τουρκίας μηνιαίως, γύρω στα 25 ευρώ. Και με αυτή την κάρτα λοιπόν την πιστοτική οι πρόσφυγες μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους και τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ σε κάποια συμβεβλημένα καταστήματα. Τους επιτρέπεται επίσης να εργαστούν οι πρόσφυγες σε κάποιες τουρκικέ επιχειρήσεις. Ήδη συμβαίνει αυτό. Υπάρχει παράλληλη οικονομία η οποία αντιπροσωπεύει γύρω στο 40% του χώριου προϊόντος της Τουρκίας. 25 στρατόπεδα λοιπόν που φιλοξενούν συνολικά 250.000 πρόσφυγες 90 όμως της 100 των Σύριων προσφύγων ζουν εκτός στρατοπέδων επειδή ακριβώς δεν... και ζουν μάλιστα συνθήκες οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε γύρω στις 800.000 παιδιά από τη Συρία και τρακόσια μόνο παιδιά έχουν πάει στο σχολείο, 300.000 παιδιά από αυτές τις 800.000 έχουν πάει μόνο στο σχολείο, οπότε εδώ διατρέχουμε το κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς. Με τις επιπτώσεις που μπορείτε να φανταστείτε. Η Ευρώπη λοιπόν αντέδρασε. Θα θυμάστε είχαμε την ανακοίνωση του Νοέμβρη για τη Συρία, όταν είχαμε ψηφίσει δηλαδή τον ε, προπολογισμό του 16 χωρίς να ξέρουμε τότε ακριβώς ε, πώς θα χρηματοδοτούσουμε αυτές τις δράσεις μας, πάντως είδαμε ότι κάποια κονδύλια, κάποιες πιστώσεις οι οποίες προέρχονταν από το εργαλείο της προσχώρησης που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ε, στην περίοδο 7-13, κάποια λοιπόν από αυτά τα κονδύλια και πιστώσεις μας ε, επέτρεψαν να τις χρησιμοποιήσουμε περίπου σε ύψος ενός δισεκατομμυρίου. Βεβαίω εξαρτάται και από τη συμμετοχή των χωρών μελών, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια συμβάλλει με ένα ποσό τη τάξης των 250 εκατομμύριων ευρώ. Ανακοινώθηκε λοιπόν μια υποδομή για τους πρόσφυγες στην Τουρκία που θα περιλαμβάνει κονδύλια 3 δις ευρώ και το ένα δίστα προέρχεται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και με αγωνία θα δούμε ακριβώς το πώς θα βρούμε τα κονδύλια αυτά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένω για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, το θέμα είναι να δούμε ακριβώ τι κάνει η Ευρώπη σε συνθήκε ακριβώ τόσο δραματικέ, με διακυβεύματα τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε λοιπόν ε, την εκπαίδευση, την παιδεία των παιδιών αυτών και πρέπει να δούμε πώς θα τα πούμε όλα αυτά όταν συναντάμε ας πούμε άτομα όπως τον κύριο Σιμψέκ, ε, υπουργό παιδείας που είναι και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, λέγοντας ότι κοιτάξτε εδώ και να χάσουμε χρόνο και ότι οι Τούρκοι από τώρα θα πρέπει να ανακοινώσουν και να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους. Και να του πούμε ότι κοιτάξτε μην χάνετε χρόνο εδώ, υπάρχουν οργανισμοί ε, που έχουν τεχνογνωσία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκόσμια Τράπεζα. Γιατί λοιπόν να μην εμπιστευτούμε αυτού του εμπειρογνώμονε, αυτού του ειδήμονε, ακριβώ για να κάνουμε μια αξιολόγηση των διαφορών προγραμμάτων και να κινητοποιήσουμε τάχιστα τα κονδύλια. Φαίνεται όμω ότι οι διαδικασίε δεν είναι και τόσο απλέ. Υπάρχει περιπλοκότητα, υπάρχει αδράνεια και το είδαμε σε διάφορα προγράμματα Γίνονται έτσι κάποιες ανακοινώσεις, αλλά τέλος πάντων δεν φτάνουν στο τελικό προορισμό αυτές οι προσπάθειες. Και υπάρχει και κάποια καχυποψία. Πώς μπορούμε λοιπόν να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και Τουρκίας. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το ζητήσαμε αυτό από τις ε, τουρκικές αρχές, να είναι όσο πιο διαφανής γίνεται σε επίπεδο κυβερνήσεις αλλά και σε επίπεδο συλλογικοτήτων γιατί ας πούμε στις πόλεις της Νότιας Τουρκίας ο πληθυσμός των προσφύγων είναι μεγαλύτερος από τους αυτόχθονες, από τον αυτόχθονα πληθυσμό. Φαντάστε λοιπόν τι επιπτώσεις υπάρχουν σε επίπεδο υγιεινή, σε επίπεδο εκπαίδευση των παιδιών, προβλήματα δηλαδή τα οποία πρέπει να λυθούν και τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Οπότε, πώς να επεκτείνουμε τη βοήθειά μας σε αυτούς που ζουν εκτός στρατοπέδων. Η UNICEF έχει λάβει μια πρωτοβουλία για να χτιστούν κάποια σχολεία και να αναλάβει τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας των δασκάλων σε συνεργασία βέβαια με τις εθνικές και τις ε, τοπικές αρχές. Τώρα πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην εργασία αυτών των ατόμων χωρίς να δημιουργηθούν συνθήκες άκρας ανταγωνιστικότητας, οι οποίες θα μπορούσαν τέλο πάντων να δυσκολέψουν τις ε, βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες ε, σήμερα πρωταγωνιστούν στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Όταν λοιπόν λάβαμε την απόφαση να επεκτείνουμε την Ευρωπαϊκή, μάλλον την Τελωνιακή Ένωση προς την ε, Τουρκία, κατά κάποιο τρόπο δευκολύναμε τη μετεγκατάσταση διαφορών ε, δραστηριοτήτων από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Και σήμερα η Τουρκία σε οικονομικό επίπεδο στην ουσία μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε ένας από αυτού τους συνομιλητές συμφώνησε μαζί μας ότι πραγματικά το βαθύ πρόβλημα, μάλλον τα βαθιά αίτια του προβλήματος των προσφύγων στην Ευρώπη βρίσκονται στη Συρία όπου η επικαιρότητα πραγματικά μας παρουσιάζει διάφορες στρατιωτικές επιβάσεις εκ μέρους του Συριακού καθεστώτους και των Ρώσων βεβαίως, Συναντήσαμε και στο Καζιαντέπ ένα συνομιλητή σε ένα πυρήνο ο οποίος ε, βρίσκεται υπό την ε, ευρωπαϊκή έτσι, εποπτεία Εκεί ταυτόχρονα βλέπουμε να συνεπάρχουν υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εκπρόσωποι των διαφόρων χωρών μελών της Ένωσης, οι οποίοι παρεμβαίνουν ακριβώς και είναι ενεργοί στην περιοχή του Καζιαντέπ. Και ακριβώς κινητοποιήθηκαν λόγω ακριβώς της στρατηγικής επέμβασης στο, στην Αλέπο και στο, στην Βόρεια Συρία. Το 2011 όταν τα δραματικά συμβάντα ξεκίνησαν, είχαμε 22 εκατομμύρια κατοίκους στην χώρα αυτή στη Συρία. 2 εκατομμύρια έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρει που είναι. 5-6 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, Ιορδανία, Λίβανος, Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Έχουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια τα οποία υποστηρίζουν το καθεστώς του Ασάντ και έχουμε 8 με 10 εκατομμύρια ατόμων τα οποία έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό της χώρας και λόγω των στρατιωτικών παρεμβάσεων και του καθεστώτος και των Ρώσων στο, στην Αλέπου και στο βορρά της χώρας υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ατόμων που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με την Τουρκία και τα οποία έχουν κλείσει εδώ και δύο εβδομάδες και προσπαθούν από την πλευρά των συνόρων της Συρίας στα σύνορα με την Τουρκία να στήσουν στρατόπεδα με ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση εκεί η οποία σύντομα θα είναι εκρηκτική και διαχείριστη. Έχουμε και τους δρόσους που προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να δυσκολέψουν τους Ευρωπαίους αν αυτό είναι τώρα αντίβαρο αυτό που συμβαίνει στην ε, Ουκρανία και στην Κερμαία δεν ξέρω. Πάντως η κατάσταση έχει γίνει πολύ επικίνδυνη και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μάθουν και να γνωρίζουν το μέρος που θα λάβουν όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων στο εσωτερικό της Συρίας. Φύγαμε λοιπόν με πολλές ανησυχίες και ερωτηματικά ομολόγω. Επειδή οι αρχές της Τουρκίας μας διαβεβαίωσαν ότι θα κάνουν όλα τα απαραίτητα για να μπορεί να υπάρξει και ένα είδος φράγματος μεταξύ των τουρκικών ακτών και των ελληνικών νησιών για να μπορέσουν να σταματήσουν το ρεύμα προσφύγων από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για κάποιο είδος <clears throat> φράγμα που μπορούν να <clears throat> δημιουργήσουν, αλλά φυσικά η αιτία του προβλήματος είναι η αστάθεια στη Συρία και εκεί το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την αστάθεια και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα. Αυτά λοιπόν οι κάποιες εμπειρίες που θέλησα να σας φέρω. Θέλω να υπογραμμίσω την ε, καλή οργάνωση αυτής της ε, αποστολής και να εκφράσω τη βαθιά, τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την γραμματεία της Επιτροπής μας, κυρίως προς τον κ. Μαρέ, ο οποίος προετοίμασε με μεγάλη φροντίδα αυτή την αποστολή. Θα οριστικοποιήσουμε λοιπόν την έκθεσή μας για αυτή την αποστολή. Συγχρόνως ήταν παρόντες και οι συναδελφοί μας από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε μαζί τους ενδεχομένως για να έχουμε μια κοινή έκθεση αλλά από πολλές απόψεις πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη φαίνεται αυτή τη στιγμή να αδρανεί ή τουλάχιστον καθυστερούμε πολύ να αντιδράσουμε και δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να λύσουμε τα κέρια αυτά θέματα τα οποία αναδύονται στην Τουρκία και τη Συρία. Και τώρα να στραφώ προς τους συναδέλφους που ήταν παρόντες στην αποστολή αυτή να μας πούν ποια ήταν τα, ειδικέ τους ε, εμπειρίες και εντυπώσεις. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πάρα πολλά να πω, διότι η εισαγωγή σας ήταν πολύ πλήρης. Η προσωπική μου στάση ήταν ότι βρήκα εξαιρετικό το πώς η Τουρκία αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά όταν σκέφτομαι την ιστερική συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη. Θυμάμαι τον κύριο που μας μίλησε για χειρονομίες. Ε, μας μίλησε για τους ε, ε, φιλοξενούμενους. Μας είπε ότι είναι δώρο του Θεού ο προσκεκλημένος. Φανταστείτε στη Γερμανία να μιλάνε για κάτι τέτοιο. Έχουμε, έχουν 2,7 εκατομμύρια πρόσφυγες στη χώρα τους. Η Ομοσπονδιακή Γερμανία έχει λιγότερο από τους μισούς. Ε, τίθεται το θέμα αν τους βλέπει κανείς σαν βάρος ε, ή σαν ε, ευκαιρία και βρίσκω αξιοθαύμαστο αυτό που έχει κάνει η Τουρκία. Η τουρκική πλευρά επιχειρηματολογεί ότι μέχρι τώρα 9 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια έχει δαπανίσει για να καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση όσον αφορά τους πρόσφυγες. Και θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια τη συζήτηση για την απελπιστική κατάσταση του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων που μίλησε για τα κύματα προσφύγων προς την Ευρώπη. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τώρα το πρόγραμμα αυτό ε, χρηματοδοτείται πιο καλά από ό,τι πέρσι, αλλά 50 τουρκικές λίρες ε, το άτομο αναμίνα μήνα αρκούν για να μην πεθάνει κανείς από την πείνα. Για να βοηθήσουμε λοιπόν το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, πιστεύω ότι είναι αυτονόητο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αφήσει τους ανθρώπους αυτούς εκεί που είναι, κοντά στην πατρίδα τους ε, και να... προλάβουμε απελπιστική κατάσταση όσον αφορά τα τρόφιμα, κάτι που θα τους οδηγήσει προς την Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, τα νούμερα της UNICEF, 310.000 ε, παιδιά πάνε σχολείο στα σχολεία της ε, UNICEF ε, στην Τουρκία. Πάνω από 100.000 παιδιά το χρειάζονται αυτό όμως. τον πολιτικό αυτό στόχο δεν θα πρέπει να τον αποφύγει η Ευρώπη. Εάν μπορεί να φροντίσει τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν σχολείο κοντά στην πατρίδα τους ε, και να διδάσκονται από Σύριους δασκάλους, θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Σκεφτείτε άλλωστε τις ε, δημοτικές υποδομές, ε, για παράδειγμα την αποκομιδή απορριμμάτων και λοιπά στις περιοχές όπου φτάνουν οι Σύριοι πρόσφυγες. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες και να φροντίσουμε η βοήθεια να καταφτάνει στα σημεία όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη. Και δεν θέλω να αμφισβητήσω την εμπειρογνωμοσύνη της ε, Ευρώπης, αλλά η σκέψη να χρησιμοποιήσουμε το ευρωπαϊκό χρήμα ως μόχλευση αυτό θα πρέπει να μου το εξηγήσει κανείς προτού να ακολουθήσω αυτήν την πολιτική σκέψη, διότι νομίζω ότι οι άμεσες ε, επιδοτήσεις είναι ο δρόμος που θα πρέπει να εξερευνήσουμε. Από τις πολλές ε, συζητήσεις που είχαμε, εγώ πρόσεξα ιδιαίτερα το εξής. θα ήθελα να προσέξω ιδιαίτερα και να ρωτήσω την Κομισιόν οι χρηματοδοτικές ροές. προς την Τουρκία ε, Πώ τις έχει φανταστεί, δηλαδή σε ποιο ταμείο πάνε. Για παράδειγμα, όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, μπορεί κανεί ε, να μεταφέρει ε, άμεσα τα χρήματα προς την UNICEF, ε, προς τους Δήμους της Τουρκίας, όμως ξαφνικά δυσκολεύει η κατάσταση. Πώς λοιπόν ε, θα πραγματοποιηθεί αυτή η ροή χρημάτων. Και θα υπάρχει κάποιο τέλος διαχείρισης ε, των χρημάτων αυτών, διότι υπήρχε η σκέψη να Υπάρχουν προσπάθειες για τα σχολεία, για τα τρόφιμα κλπ. Μπορούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές. Ε, εγώ θα ήθελα όμως ε, τα χρήματα που δίνει η Ευρώπη ή τα κράτη-μέλη να γνωρίζω ότι καταφτάνουν, ε, ότι τα παίρνουν τελικά οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Και θα ήθελα να δω μια σχετική πιστική απάντηση γι' αυτό. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να συντομεύσουμε λιγάκι. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, κύριε Ρούμπιχ. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Η παρουσίασή σας έδειξε πολύ καθαρά ότι εδώ έχουμε μία σημαντική σύγκρουση της εξωτερικής πολιτικής, όχι αμάνεστα στους Σουνίτες και τους ε, Σιήτες, οι ΣΥΤΕ στηρίζονται από το Ιράν και την ε, Ρωσία, οι ε, άλλοι από την Αμερική και του άλλους. Από την άλλη έχουμε και τη σύγκρουση με τους Κούρδους. Ε, η Τουρκία βρίσκεται εν μέσω μιας πολλαπλής σύγκρουσης και θα πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Και αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι και ο Ασάντ έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε υπολογίζουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα καταφτάσουν 400 με 600 χιλιάδες πρόσφυγες στα τουρκικά σύνορα και πρόκειται για αριθμό ανθρώπων που θα παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα, διότι τα σύνορα προς την Τουρκία παραμένουν λίγο πολύ κλειστά. Θα βρεθούν λοιπόν κάπου ανάμεσα στη Συρία και στην Τουρκία. Η βοήθεια των διεθνών οργανισμών χορηγείται με εντατικούς ρυθμούς. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πρόσφυγες στα σύνορα της, Τουρκίας, της Συρίας να λάβουν όσο γίνεται καλύτερη βοήθεια. Η Τουρκία ανα πρόσφυγα δίνει 30 λίρες το μήνα. Εμείς ε, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τέτοιες δράσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, τι ζητάνε για να κάνουν κάτι τέτοιο. 3 με 18% είναι οι παρακρατήσει των μη κυβερνητικών οργανισμών. Τι ακριβώ καλύπτουν αυτέ. Θέλουμε η βοήθεια να φτάσει σε αυτού που την έχουν ανάγκη. Τι μέσα έχει στη διάθεσή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξει την κατάσταση. Είδαμε ότι οι Τούρκοι διαθέτουν τρόφιμα, φάρμακα με αποτελεσματικό τρόπο, παιδεία, ιδιαίτερα διδασκαλία της γλώσσας. Παρ' όλα αυτά έχουν πάνω από 20 καταβλισμούς με 10.000 πρόσφυγες ο καθένας, οι οποίοι σίγουρα χρειάζονται βελτίωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε οι άνθρωποι να παραμείνουν όσο γίνεται πιο κοντά στις πατρίδες τους. Ελπίζουμε σύντομα να, υπάρξει, να επικρατήσει πάλι η ειρήνη. Άλλωστε πολλοί από τους πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Τουρκία με τα αυτοκίνητά τους. Είναι καθήκον των διεθνών οργανισμών, για παράδειγμα του ΟΗΕ, να ε, δημιουργήσει εκεί μια ε, ζώνη με κιανόκρανους για να προστατεύσει τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέργκερ. Μια μικρή προσθήκη και αίτηση κύριε Πρόεδρε. Το τελευταίο μήνα εμείς έχουμε ζητήσει από την Κομισιό να μας δώσει πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται η πληρωμή όλων αυτών των ταμείων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης και το τι γίνεται με το παγκόσμιο προ... πρόγραμμα τροφίμων. Και προφανώς περιμένουμε ότι θα αυξηθούν οι απαιτήσει στον τομέα αυτό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο η Κομισιόν να μας δώσει το ταχύτερο να το μια συνολική επισκόπηση για να μπορούμε να έχουμε μια αξιολόγηση για την ε, και τα αριθμητικά ποσά με τα οποία εργαζόμαστε και να έχουμε μια αξιολόγηση <clears throat> και επίσης να δούμε τι γίνεται με αυτά τα οποία φασίστηκαν στην συνεδρίαση των ε, δωρητών στο Λονδίνο και τα ποσά τα οποία έχουν υποσχεθεί όλοι αυτοί δεν έχουν ακόμα φτάσει εκεί. Δεν πρέπει λοιπόν να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όπως τα προηγούμενα χρόνια που έρχονται όλα κατόπιν εορτής θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μήνα έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα του πώς εξελίσσεται η κατάσταση, αν έχει αρκετά κονδύλια ακόμα το πρόγραμμα του ΟΗΕ για, για τα τρόφιμα και πώς αντιμετωπίζεται το θέμα των ε, προσφύγων, γιατί μπορεί να προκύψουν καταστάσεις που αλλιώς δεν θα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε καθόλου. Για το εκατομμύριο του καταπιστεύματος το δισεκατομμύριο για το καταπίστευμα της Συρίας, νομίζω 40% έχει εκταμιευτεί αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δείχνει πόσο βραδιπορεί το σύστημα. Οι διαδικασίες, ο συντονισμός, όλα αυτά. Είναι σαν να έχουμε μια πυρκαγιά και οι πυροσβέστες συζητάνε για το πόσο κοστίζει το λίτρο του νερού για να ξέρουν αν θα κάνουν ή όχι μια ενέργεια πυρόσβεσης. Ο κύριος Σομαζέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <coughs> γυρίζοντας από αυτή την αποστολή, νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγα λεφτά να σας δώσω την συνολική μου εντύπωση. Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα τα οποία βρήκαμε ενώπιόν μας. Εγώ γυρίζω όμως με την βεβαιότητα ότι, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια απλοϊκή απάντηση σε προβλήματα τα οποία είναι εξόχως πολύπλοκα. Αυτό ήταν ένα ταξίδι στο κέντρο, στον πυρήνα της πολυπλοκότητας της Μέσης Ανατολής, Μέση Ανατολής που τώρα έχει πραγματικά γίνει ακόμα πιο πολύπλοκη και επίσης είναι και ένα μάθημα πολυπλοκότητος για την κατάσταση στην Τουρκία και για τον αντίκτυπο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τις τρεις αυτές λοιπόν πτυχές χρειάστηκε να τις αντιμετωπίσουμε στο ταξίδι μας. Ποια είναι δική μου εντύπωση μετά από την ε, επίσκεψη στον καταβλισμό στο Οσμανιγέ. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο για μας ως ευρωβουλευτές να μπορούμε να δίνουμε μαθήματα σε ένα κράτος σε σχέση με τις συνδίκες υποδοχής των προσφύγων. Τόσο ανάξιοι είμαστε, όσο είμαστε εμείς τόσο ανάξιοι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να δώσουμε μια σωστή απάντηση στην υποδοχή των προσφύγων. Και εγώ ως Γάλλος, αν σας θυμίσω τι συμβαίνει στους καταβλισμούς στο Καλέ που δεν ανταποκρίνονται σε κανένα πρότυπο και προδιαγραφή, νομίζω ότι ενώπιον των Τούρκων, παρά το γεγονός ότι είχα πολλά ερωτήματα, προτίμησα να σιωπήσω. Το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, μας είπαν οι Τούρκοι ότι έχουν δαπανίσει περίπου 9 με 10 <clears throat> εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων. Θα πρέπει τώρα να δούμε κατά πόσο μπορούμε να διακριβώσουμε αν είναι σωστά αυτά τα στοιχεία ή όχι. Αυτό όμως το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι αυτή η χώρα σήμερα υποδέχεται πάνω από 2,7 εκατομμύρια προσφύγων, ενώ στην Ευρώπη έχουμε τεράστιες δυσκολίες να πράξουμε κάτι αντίστοιχο. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν τι θα σήμαινε για τις κοινωνίες μας να έχουμε ένα τέτοιο αριθμό προσφύγων και πόσο πιο δύσκολα ακόμα είναι τα πράγματα αυτά για την Τουρκία. Και υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση. Εγώ γυρίζω με την εικόνα ότι πίσω από αυτό το, τη γενική έννοια του, του πρόσφυγα υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν οικογένειες, έχουν προσωπικό ιστορικό, έχουν μια ζωή που έχουν αφήσει και δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε μέσα στην πολιτική που ακολουθούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν η αντιπροσωπεία μας να συζητήσει και με την ε, αποστολή της Λίβε που ήταν παράλληλα με μας στην Τουρκία για να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα το κάνουμε λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, μένουμε σε αυτό το επίπεδο. Εάν δεν έχετε αντίδυση θα επανέλθουμε. Αυτό το οποίο είδαμε βέβαια είναι να, υπάρξει, να υπάρχει μια έλλειψη ηγεσία. Υπήρξε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων που εμπλέκονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτοπίως και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα θα πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο. Θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μπορεί να έχει μια ηγετική θέση στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα τώρα το οποίο τίθεται είναι πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τις, ε, τα αιτήματα των τουρκικών αρχών, επίσης τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέω για τον κύριο Γιάρα αυτά που μας είπε ο κύριος Σιμσεκ δεν είναι για να γίνει μια έκκληση στην Παγκόσμια Τράπεζα ή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τα Τρόφιμα. Ουσιαστικά το θέμα είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη τους ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε με οκίτητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Συρία έχουμε χιλιάδες άτομα τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη απόγνωση. Εάν δεν υπάρξει σωτηρία για τα άτομα αυτά, ο κίνδυνος ρίζος παστικοποίησης, γιατί είναι πολύ παρούσα, είναι παρόν πράγματι και το Ισλαμικό κράτος στη Βόρεια Συρία, ο κίνδυνος είναι να οδηγηθούν τα άτομα αυτά στην ριζοσπαστικοποίηση και μπορούμε να φανταστούμε τι θα σημαίνει αυτό σε γεωπολιτικό επίπεδο και ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω λοιπόν αυτά τον απολογισμό της αποστολής μας που ήταν τόσο ενδιαφέρουσα και καλά οργανωμένη και ευχαριστώ την γραμματεία και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μούρεσαν για την έκθεση για την ε, αηφόρο ε, εταιρική σχέση αλίας με τη Λιβερία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομοδότηση της Επιτροπής μας μετά την έκθεση της Επιτροπής Αλίας, δύο λεπτάκια μόνο. Έχουμε μια συμφωνία λοιπόν αλίας μεταξύ της Ένωσης και της Λιβερίας που προσπογράφηκε στις 15 Ιούνιου πέρσι. Στόχος είναι να δοθούν στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ευκαιρίες και το δικαίωμα αλλιεύσης στα ύδατα της Λιβερίας. Για τα είδη τόνου και τον ίδιο τον τόνο. Παρόμοιε συμφωνίε έχουμε με άλλε Αφρικανικέ χώρε, μεικτέ συμφωνίε. Η επιδόση τώρα για τον προπολογισμό τη Ένωση. Χρειαζόμαστε 25.000 ευρώ για τον πρώτο γεωσυμφωνία, 600 για το δεύτερο έτος και 580 δηλαδή γύρω στα 3,5 κάπου εκατομμύρια ευρώ από τον προπολογισμό μας για τη χρηματοδότηση αυτής, χρηματοδότηση αυτής της συμφωνίας αλληλείας με την Λιβερία που είναι πενταετής. Καταρχάς αυτό για να στηρίξουμε τις αρχές πολιτικές της ε, Λιβερίας για τον ε, έλεγχο και την εποπτεία. Μετά το τονάς και η αναφορά 650.000 του ετησίως. Αν αλεύσουμε περισσότερο, τότε η χρηματοδοτική εισφορά θα είναι 55 ευρώ ανατόνο το πρώτο έτος, 50 το ανατόνο το δεύτερο και τρίτο έτος και 45 ευρώ το τέταρτο και πέμπτο έτος. Επειδή λοιπόν αυτή η συμφωνία δεν είναι προβληματική, σας προτείνω να υιοθετήσουμε αυτή τη συμφωνία και να καλέσουμε την Επιτροπή Αλίας ως αρμόδια να μας υποβάλει θετική πρόταση και οι προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι 24 του Φλεβάρη. Στη συνέχεια θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας στις 16-17 Μαρτίου και η ψηφοφορία της έκθεσης της Επιτροπής Αλίας θα γίνει κατά διάρκεια της Ολομέλειας του Απρίλη φέτος. Αυτά προεδρευομένα. Ευχαριστώ πολύ. Pardon. La parole. Ευχαριστώ κυρία Καθαρτάμπαλ για την έκθεσή της Αλία μεταξύ, συμφωνία Λύσης μεταξύ Ένωσης και Μαυρτανίας. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Όπως είπαμε, μιλάμε για την ανανέωση του πρωτοκόλου συμφωνίας αλίας μεταξύ Μαυριτανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ως Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να εγκρίνουμε το χρηματοοικονομικό κομμάτι, 59 εκατομμύρια το έτος, 55 για τα αλλιεύματα και 4 εκατομμύρια τα οποία αφορούν τεχνική συνεργασία, επιστημονική συνεργασία, κατάρτιση, προστασία περιβάλλοντος κλπ. κλπ. Να πω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη συμφωνία τούτη, οπότε ζητώ θετική ψήφο για αυτή την ε, συμφωνία και ανανέωση αυτού του πρωτοκόλλου που Νομίζω θα ψηφίσουμε το Μάρτιο εδώ στη δικιά μας την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις, ρωτάει το Πρόεδρος. Όχι από ό,τι βλέπω. Να σας πω τότε ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 24 του Φλεβάρι και ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα γίνει στις 16 ή 17 Μαρτίου. θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σας καλώ να βάλετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες στο μηχάνημα μπροστά σας, ώστε να μπορέσουμε, αν χρειαστεί, να ελέξουμε και να ψηφίσουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία, επιτρέψτε μου να πω, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ που ψηφίσατε. 24 κάρτες μπήκαν. 21 ψήφους έχουμε μέχρι τώρα. Κύριε Γκάγερ, έχετε ψηφίσει. Εντάξει. Ωραία. Αποφασίζουμε λοιπόν για την έκθεση η οποία αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Να σας πω προς την κυρία Βάνα κυρίως, ότι ως Πρόεδρος είχα κηρύξει μη αποδεκτή διακόπτη ο Πρόεδρος. Είχα, κύριε, είχα χαρακτηρίσει μη αποδεκτή την 30 30η τροπολογία αλλά το αποσύρω αυτό. Οπότε σας καλώ να ψηφίσουμε για τροπολογία τούτη της κυρίας Βάνα, την παρθμό 31. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. <coughs> Απορρίπτεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μπε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με δύο τροποποιήσεις υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 15-10. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. <coughs> Εγκρίνεται. 18. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 με χωριστή ψηφοφορία για τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά ψήφι υπέρ κατά αποχές. Δεν σηκώσατε όλοι τα χέρια. Ζητώ να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 19-5 με μια αποχή. Το υπόλοιπο λοιπόν στις 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 14-11. Συμβαστική σε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπάρχουν όμως, συγγνώμη, υπάρχουν ψηφοφορίες για ορισμένα τμήματα τα οποία είναι κίτρινα. Η δεύτερη παύλα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτη παύλα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτη παύλα υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Τέταρτη παύλα άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 14-11 Απολογία 30 τώρα. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την 31. Πέρασε. 14-9 απορρίπτεται με δύο αποχές. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15-9 απορρίπτεται. Το σύνολο τώρα του κειμένου πως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκαεπτά εναντί οκτώ με καμία αποχή. Και ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση του Τωμά Ζεστόφσκι για την αλληλευτική συμφωνία με την Γερμανία και την Γρυλανδία. Υπάρχει μία μοναχα ψηφοφορία, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ονομαστική κλίση, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο ψηφοφορίες. Ψήφι υπέρ. Δανία. Αλία. Με τη Δανία και τη Γερλανδία. Λοιπόν, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υποστηρίχθηκε λοιπόν η συμφωνία για τη γνωμοδότηση τώρα. Πάλι μονομαστική κλίση. Μονομαστική κλίση τώρα μάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Μία και μία αποχή. άλλα τμήματα του προϋπολογισμού με τον κύριο Ντεπρέ, τροποποίηση του οργανογράμματος, μόνο για μία θέση στο οργανόγραμμα. 10 Φεβρουαρίου είχαμε πάρει ειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ότι θα τροποποιήσει βάσει του άρθρου 50 του Δημοσιονομικού Κανονισμού το οργανόγραμμά του, ε, απεστάλλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού η πρώτη τροποποίηση του οργανογράμματος βάσει του άρθρου 51 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και παρουσιάζεται για πληροφόρηση σε εμά. Είναι μια θέση μονάχα και εάν τα λέω σωστά, όπως λέει ο κ. Δεπρέ, δεν χρειάζεται να υπάρξει κάποια παρατήρηση από τη δική μας πλευρά. Μπορεί να γίνει δεκτή λοιπόν αυτή η αίτηση ως έχει, δεν έχουμε καμία αίτηση για την κτηριακή πολιτική. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε κλείσει την συνεδρίασή μας. Υπάρχουν άλλα θέματα. Όχι. Λήξη της συνεδρίασης. Επόμενη συνεδρίαση 18 Φεβρουαρίου την 5η το πρωί από τις 9 ως τις 12.30. Και τώρα θα ακολουθήσει η έκτακτη και επίσης θα υπάρχει στις 23 Φεβρουαρίου μια έκτακτη συνεδρίαση εδώ στις Βρυξέλλες. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών.